Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω υπόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξαιρετικά περιστατικά και εξελίξεις που έχουμε στην γαλλική δημοκρατία, που πλήττουν ε, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου. Ε, πρόκειται για παραβίαση των ε, προσωπικών ελευθεριών. Πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην υπουργοί και νομικοί υπέστησαν παρακολουθήσεις ε, των ε, τηλεφωνικών τους ε, συνομιλιών. Πρόκειται για μια παράδεκτη κίνηση κατά της προσωπικής ελευθερίας και της δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 7 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναφέρει ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα σεβασμού της προσωπικής του ζωής όταν ε, ψηφίσαμε την έκθεση Μωραές για τις ε, υποκλοπές της NSA ε, ζητώ μήπως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε αυτές τις εξελίξεις στην Γαλλία μήπως θα μπορούσαμε να κινήσουμε τη διαδικασία παραβάση. Ευχαριστώ κύριε Μποντή. Έχω ενημερώσει τους αρμόδιους. Ξεκινάμε λοιπόν ε, την ψηφορία. Ξεκινάμε την έκθεση Σάλα. Μία ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται.